Hello. Εμπρός. Εμπρός με ακούτε. Ναι, ναι, σας ακούμε κύριε Λόπες Αγγελάου. Όπως προείπαμε, πρέπει να κάνουμε μια ψηφοφορία με την ίδια διαδικασία. Σύμφωνα με κάποια λίστα, να στείλετε την ψήφο σας στη γνωστή διεύθυνση email. Συν πλην μηδέν είναι η αποχή σε το την ειδική διεύθυνση email για να μετρήσει ψήφο και στις 4 η θα έχουμε ανακοινώσει τα αποτελέσματα τη ψηφοφορία. Καλώ. Εντάξει, με ακούσατε. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα προχωρούμε. Πάμε τώρα στα σημεία ουσίας της σημερινής συνεδρίασης, αλλά να ληφθεί υπόψη Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό, διακόπτεται. Να δούμε αν έχουμε απαρτία. βεβαίω, βεβαίω, να δούμε αν έχουμε απαρτία. Παρακαλώ, πιέστε το σχετικό κουμπί για να δούμε αν έχουμε απαρτία. Είναι θέμα διαδικαστικό. Καλώς. Ας μου πει η γραμματεία, αν υπάρχει απαρτία, μάλιστα υπάρχει, σας το επιβεβαιώνουμε. Οπότε πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της μέσας διάταξης, το θέμα ουσίας, όσον αφορά την εκτίμηση ε, ενός σοβαρού κινδύνου για παραβίαση των διατάξεων σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία. Κύριε Θαρταλέχος, κύριε Θαρταλέχος, Μα ακούτε? Έχουμε στην του κύριο Θαρθαλέχο. Θέλατε κάποιο διαδικαστικό. Θαρθαλέχο. Ναι, ναι, ναι. Ήθελα το λόγο, ναι. Και σας ακούω. Έχετε ένα λεπτό του, λέει ο Πρόεδρος. Και διακόπτεται η σύνδεση. Θαρθαλέχος. Ο Ρουίς έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία του Καβαγέρο στην Παμπλώνα. Είναι μέλος αδελφού κόμματος του Λαϊκού Κόμματος. Είχαμε 853 θύματα της ΕΤΑ και για τη δολοφονία αυτών δεν έχει καταδικαστεί Κανείς. Κανείς δεν χαρακτήριζε αυτόν τον άνθρωπο ως ε, ένοχο ανθρωποκτονίας και θεωρείται πολιτικός κρατούμενος. Εμείς θέλουμε να σας πούμε ότι θα πρέπει να μην θεωρούμε πολιτικούς κρατουμένους αυτούς που είναι κοινή δολοφόνια. Ο Πάτσι Λουίς είναι ένας ένοχος ανθρωποκτονίας δεν είναι καθόλου πολιτικός κρατούμενος. Καλά, τώρα μας το λέει ο Πρόεδρος, μας είπατε αυτό το οποίο θέλατε, κάτι το οποίο έχει σχέση με προηγούμενες με τις διάταξεις. Οπότε, ας προχωρήσουμε και πάμε στο σημείο υπαριθμών 8. Αξιολόγηση του σαφούς κινδύνου όσον αφορά την σοβαρή παραβίαση του κράτους δικαίου στην ε, Πολωνία. Έχουμε εδώ κάποια έκθεση που έχω αναλάβει και έχουμε και κάποια γνωμοδότηση για το ζήτημα αυτό από την Επιτροπή Γυναικών. Η συγγήτρια είναι η Εβελίν Ρέγνερ, η πρόεδρος της Επιτροπής των Γυναικών και έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Χωσέ Γκρέχα Μάτος που είναι ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών. Επίσης θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με την ε, κυρία Γιωχάνα Ετνάροβιτ Σίκορα μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ένωση Πολωνών Δικαστών με την ε, ονομία Γιουστίτσια. Οπότε ας προχωρήσουμε σε μια τέτοια ανταλλαγή απόψεων πριν δούμε ε, για τις ε, εξελίξεις που αφορούν το κείμενό μας, για το τι έχει γίνει πρόσφατα στη χώρα. Έχουμε καλλιτέχνες που διαμαρτύρονται και είχαμε για επιβολή προστίμου 2.200 ευρώ, διότι θεωρήθηκε ότι υπάρχει παραβίαση ε, δημιουργικών κανονισμών. Επίσης, ε, ο διαμεσολαβητής της χώρας προσέφηκε στο ε, διοικητικό δικαστήριο τη χώρα όσον αφορά μια παραβίαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα. Έχουμε επίση κάποια πειθαρχικά μέτρα κατά των ε, δικαστών που προσέφυγαν στο Δικαστήριο ε, ε, Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων και επίσης το κρατικό δίκτυο, ραδιοφωνικό δίκτυο Τρόικα κατηγορήθηκε μέσα εβδομάδα ότι ε, λογόκρινα ε, τον κατάλογο με τις μουσικές ε, επιτυχίες. Και επίσης ε, έβαλε κατά του ε, κατά, κατά, κατά κάποιου τραγουδιού που ήταν κατά του Προέδρου Κατσίνσκι. Και έχουμε τώρα επομένως μια έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 7 της συνθήκης. Όμως, πριν παρουσιάσουμε αυτή την ενδιάμεση έκθεση, θα πρέπει να ευχηθούμε να το καλωσόρισαν οι καλεσμένοι μας. Έχει ο Χωσέ πρώτος το λόγο για 7-8 λεπτά, όχι περισσότερο, ε, και κατόπιν θα υπάρξουν ερωταπαντήσεις με τους συντονιστές. Οπότε στη συνέχεια ο υποφαινόμενος θα λάβει το λόγο και θα σας ε, παρουσιάσω αυτό το κείμενο το οποίο τώρα συζητούμε που θα έχει τη μορφή εκθέσεως. Οπότε πρώτα πρώτα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ιγρέχα Μάτος, ο οποίος εκπροσωπεί την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών. Έχετε το λόγο κύριε για 7-8 λεπτά, το πολύ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας, ευχαριστώ, σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση από πλευρά τη Ενωσισμού μου και θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξαιρετική έκταση την οποία ε, καταρτήσατε. Θα μιλήσω στα αγγλικά. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω και πάλι κύριε Πρόεδρε ε, Χουάν Λόπες Αγγιλάρ με το πιο προφανή τρόπο γιατί χαιρόμαστε που επιτρέπετε στην Ένωσή μας να παρίσταται στη σημερινή συνεδρίαση να πούμε ευθύ εξ αρχής ότι είμαστε πολύ εντυπωσιασμένοι από το σχέδιο της έκθεσης. Ε, τα περιστατικά που αναφέρονται μιλούν από μόνα τους για το πώς έχει η κατάσταση σήμερα στο πολωνικό δικαστικό σώμα. Αυτό το λεπτομερές ε, ενδελαχέ έγγραφο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και σε ό,τι αφορά τα προτινόμενα μέτρα για το μέλλον ελπίζει η Ένωση Δικαστών ότι θα πετύχουμε να έχουμε μια στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικά και ειδικά με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Α εργαστούμε λοιπόν πιο, ας συνεργαστούμε πιο στενά για να προστατεύσουμε το κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών, ένα περιφερειακό τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Δικαστών που ιδρύθηκε το 1953, είναι κατά πολύ η μεγαλύτερη οργάνωση που εκπροσωπεί δικαστές στον κόσμο. Είμαστε λοιπόν, ε, συναπαρτιζόμαστε από τις κορυφαίες εθνικές ενώσεις δικαστών σε 44 χώρες, κυρίως ε, σχεδόν όλων των ε, χωρών από την Ήπειρό μας. Αυτή η μακροπρόθεσμη λειτουργία της οργάνωσής μας εξηγείται από την απόλυτη προστασία και απομόνωση από πολιτικές παρεμβάσεις. Είμαστε εντελώς μη πολιτικοί και βασική μας αποστολή είναι η ανεξαρτησία, η δικαστική ανεξαρτησία και το κράτος δικαίου. Ένας ε, δικαστής λοιπόν θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, να μην έχει, ε, να μην υπόκειται σε κανένα δασμικό όργανο, να μην δέχεται ε, εντολές, διαταγές από κανένα άλλο όργανο και να προστατεύεται από εξωτερικές ή ιστορικές πιέσεις. Αν ε, λοιπόν ένα κράτος ε, δεν ε, εγγυάται στους δικαστές του την εξαρτησία τους, δεν μπορεί να θεωρείται δικαστής ή δικαστής πλέον. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι είναι ένας εμπειρογνώμονας, ο οποίος θα έχει νομικές γνώσεις, αλλά στην τελική ανάλυση δεν θα είναι δικαστής, ο οποίος θα υπηρετεί τους πολίτες, τους συμπολίτες μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών, λοιπόν, από την πρώτη ημέρα απέρριψε τις επιθέσεις κατά της δικαστικής ανεξαρτησίας στην Πολωνία. Οι διαρκείς προειδοποιήσεις από πλευρά μας ελήφθησαν υπόψη και σε συνεργασία με άλλα διεθνή σώματα, το ENCJ, το Δίκτυο Προέδρων Ανατοτάδων Δικαστηρίων, τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για δικαστές και δικηγόρους CG κτλ. Στι 1η 11 Ιανουαρίου, λοιπόν, σε μια ιστορική στιγμή, εκατοντάδε δικαστέ από ε, δεκάδε ευρωπαϊκέ χώρε ε, διαδήλωσαν στι ε, δρόμου τη Βαρσοβία. Και χιλιάδε πολίτε βγήκαν μαζί μα και σε κάποιε περιπτώσει μέχρι και με κλάματα διαδήλωσαν υπέρ τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου. Σε μια τελική ομιλία, λοιπόν, αναφέραμε το θέμα των, ευρωπαϊκών, των Ευρωπαίων δικαστών. Εμείς ε, οι δικαστές λοιπόν ε, που υπερασπιζόμαστε καθημερινά σε κάθε δικαστήριο του κράτος δικαίου και όχι το δίκαιο των ανθρώπων δηλώνουμε ότι χωρίς δικαστική ανεξαρτησία θα χαθεί η ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, παρά α, όλες αυτές τις δράσεις, η διάβρωση του κράτους δικαίου στην Πολωνία είναι χειρότερη παραποτέ. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε διάφορες ε, δικαστικές αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί από ανεξάρτητα σώματα. Θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, καταρχάς, να προταθεί ε, η λήψη άμεσων, ενδιάμεσων προσωρινών μέτρων για την επιλογή ε, του Πρόεδρου του Ανατολικού Δικαστηρίου. Για να αποφύγουμε να βρεθούμε προτελεσμένου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια στρατηγική, μια στρατηγική μάλλον που χρησιμοποιεί η πολιτική η πολυνομική κυβέρνηση, θα πρέπει να υπάρχουν διάφορα επίπεδα στην διαδικασία επί παραβάση. Και θα πρέπει αυτό να περιοριστεί από δύο μήνες σε ένα μήνα το κατάνατο το όριο. Θα ήθελα επίση να τονίσω την εξαιρετική έκθεση της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ και να δοθούν ιδιαίτερη προσοχή σε διάφορε δράσει που υποστηρίζουμε. Για παράδειγμα, να υπάρχει ο κανονισμός για τον ε, προπολογισμό της Ένωσης προκειμένου να ληφθεί υπόψη η απόσυρση πόρων, παροχή πόρων προ τι ευρωπαϊκέ χώρε, ε, αν δεν υπάρχει σεβασμό του κράτου δικαίου, να καλήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει κατεπηγόντω διαδικασίε επιπαραβάσει σε ό,τι αφορά την νομοθεσία, σε ό,τι αφορά το Συνταγματικό Δικαστήριο και σε ό,τι αφορά προσωρινά μέτρα, να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει να ε, ανασταλούν οι δραστηριότητε του νέου σώματος και να εγγυηθούμε ότι αυτός ο ε, νόμος θα ε, ανασταλεί. Τούτων εχθέντων, οι διαδικασίε που παραβάσει και αυτά τα προσωρινά μέτρα, παρά την αξία τους που θα μπορούσαν να έχουν, δεν θα αρκέσουν για να αντιμετωπιστεί το συστημικό πρόβλημα που υπάρχει στην Πολωνία. Θα πρέπει να υποθέσουμε ότι όλοι και πιο πολλοί όλο και πιο πολλοί ηγέτε στην Κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη έχουν σταματήσει καν να υποκρίνονται ότι ακολουθούν του κανόνε τη δημοκρατία. Είναι λοιπόν ε, απαραίτητο τώρα, πιο πολύ από ποτέ, να προασπιστούμε τις θεμελιώδεις αξίες μα ε, σε ό,τι αφορά και τις πειρασμού που ε, υπάρχουν μια εποχή πανδημία. Οι Ευρωπαίοι δικαστές λοιπόν θα ήθελαν να προτείνουν να, να δουν ανάλογο επίπεδο αποφασιστικότητας όπως και στο Marshall Plan, το σχέδιο Marshall που καταρτίζεται για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Γιατί υπάρχει συγκεκριμένος κίνδυνος να υπάρχει αμα, μίμηση των όσων γίνονται στην Πολωνία και στην Ουγγαρία σε άλλες χώρες. Τα τρία δίκτυα που εκπροσωπούν του Ευρωπαίου δικαστέ το δίκτυο προέδρων του Ανώτατου Δικαστηρίου, Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Συμβουλίων για την Δικαστική και Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών, έχουν δείξει μεγάλη αποφασιστικότητα για να προασπιστούν την δικαστική ανεξαρτησία στην Πολωνία και σε μία επιστολή που έχει προσυπογραφεί από του τρει προέδρου προ τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα λόγια μα ήταν τα εξή χωρίς ανεξάρτητο δικαστικό σώμα σε όλα τα κράτη-μέλη, η Ένωση θα καταλήξει να αποτελεί έναν κοινό χώρο για τη δημοκρατία. Όπως είπε και ο Επιτροπός Didier Ρέιντερ σε προηγούμενη συνάντηση με την Επιτροπή, είναι απαραίτητο οι Ευρωπαίοι πολιτικοί να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα για να προστατεύσουν το κράτος δικαίου. Και για να παραθέσουμε και το Δάντη στην Ασία Κομμωδία, η πιο το χειρότερο μέρο στην κόλαση είναι για αυτού οι οποίοι σε περιπτώσει κρίσεω ε, διαλέγουν την ουδετερότητα. Συμμεριζόμαστε λοιπόν ε, τι ανησυχίε που εκφράζονται από την εισηγήτρια ότι θα πρέπει να μην επιτραπεί παθητική στάση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση τη πολύ σοβαρή κατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γνασιωμάτος. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας και επίσης γιατί μας είπατε την θέση ε, της ε, Ένωσης Ευρωπαϊκών Δικαστών ε, Πρόκειται όντως για κάποια ένωση δικαστών που είναι αμερόληπτη εξορισμού. Οπότε, στα αγγλικά. Προχωρούμε τώρα στο δεύτερο νομιλητή που έχουμε. Είναι η κυρία Ιωάννα Νάροβιτς Σίκορα που εκπροσωπεί τον Εθνικό Φορέα Ιουστίτσια, δηλαδή την Ένωση Πολωνών Δικαστών. Και εσείς έχετε το λόγο για 7-8 λεπτά το πολύ. Και σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Νίκο στην Ένωση Πολωνών Δικαστών, την οποία εκπροσωπώ. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα αλλά και μεγάλη ευθύνη καθώς γνωρίζω ότι μιλώ όχι μόνο εξ ονόματος 3.700 μελών της Ένωσής μας αλλά εξ ονόματος γενικά των Πολωνών δικαστών. Να σας πω πως με εντυπωσιάζει το σχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης, είναι λεπτομερές και συγκεκριμένο όσον αφορά και τα προτινόμενα μέτρα και έτσι συμφωνώ πλήρως με την θέση του προηγούμενου ομιλητού, του κυρίου Ζωζέ Ιγκρέα Συμφωνώ πλήρως με τα συμπεράσματα της ομιλίας του, τα οποία ε, υιοθετώ και εγώ. Όμως, θα ήθελα να παρουσιάσω κάποιες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, οι οποίες θεωρώ ότι δεν έχουν τονιστεί αρκετά στο σχέδιο έκθεσης. Εν τω μεταξύ θεωρώ ότι είναι ε, πραγματικά σημαντικό να αποκτήσετε μία εικόνα της ε, κατάστασης της πολωνικής ε, δικαιοσύνης. Έχουμε την πορεία αυτή που είχε γίνει στην Βαρσοβία, μία πόρια κατά της αναδιοργάνωσης των κατώτερων και ανώτατων ε, δικαστηρίων. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ατμόσφαιρα αυτής της πορείας όμως, παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν τότε, αλλά και πριν από τις 11 Ιανουαρίου, δεν καταφέραμε να αποτρέψουμε την καταστροφή της δικαιοσύνης στην Πολωνία. Στις 14 Φεβρουαρίου του Αγίου Βαλεντίνου είχαμε την λεγόμενη ε, νομοθεσία φήμοτρο που έχει ε, πάρα πολύ σοβαρές συνέπειες ε, για την δικαιοσύνη στην Πολωνία. Πρώτα απ' όλα, ο νόμος ορίζει ότι οποιονδήποτε ορίσει ο πρόεδρος της Πολωνίας είναι ειρηνοδίκης και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η νομοποίησή του και κάτι τέτοιο μετά είναι πειθαρχικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται μέχρι και με απόλυση. Μόνο το πειθαρχικό του ανωτάτου δικαστηρίου ε, μπορεί να αποκτήσει αν ένας δικαστής είναι ανεξάρτητος. Ο νόμος αυτός ε, έχει αράξει τον ορισμό του δικαστή, το άρθρο 55. Πάνω. Το άρθρο αυτό ορίζει ότι κάποιος έχει οριστεί ως δικαστής από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και έχει ορκιστεί για να θεωρείται δικαστής. Ε, πλέον αυτό δεν ισχύει ε, κατόπιν... Ε, ε, δεν χρειάζεται πλέον να έχει προταθεί κάποιος από το Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία ότι στόχο αυτό έχει να επηρεάσει την απόφαση του δικαστηρίου της 19ης Νοεμβρίου, την απόφαση του Ανωτά του δικαστηρίου της 23ης Ιανουαρίου και άλλες ε, διαδικασίες όπου ακόμα έκρεμουν και όπου έχει αμφισβητηθεί η αρμοδιότητα των νεοδιοριστέντων δικαστών κατόπιν ε, με τον νόμο Φήμοτρο αυξάνεται η υπαγωγή των δικαστών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. καθώς αυτοί πλέον κρίνονται από ένα συμβούλιο που ορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνη επιπλέον, οι γενικές συνελεύσεις χάνουν την σημαντικότερη λειτουργία τους και τώρα είναι ε, κάποια σώματα ad hoc. Η αυτοδιοίκηση της δικαιοσύνης ε, πλέον έχει ουσιαστικά καταργηθεί. Το δεύτερο θέμα είναι η τρέχουσα κατάσταση στο ανώτατο δικαστήριο. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο νόμος αυτός ε, έχει αλλάξει τους κανόνες ε, διορισμού των ε, δικαστών του ανωτάτου δικαστηρίου. Ως αποτέλεσμα της προηγούμενης μεταρρύθμισης του 2019, ο πρώτος πρόεδρος ορίζεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας από έναν κατάλογο πέντε υποψηφίων που υποβάλλει η Γενική Συνέλευση. Λόγω αυτής της αλλαγής η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να προτείνει πέντε υποψηφίους. Καθώς όμως κάθε δικαστής έχει μία ψήφο, καταλήγουμε τελικά ο τελικός κατάλογος των πέντε υποψηφίων να περιλαμβάνει αυτούς οι οποίοι συγκέντρωσαν πολλές ψήφους, αλλά και αυτούς που έλαβαν λίγες. Το προηγούμενο Σάββατο είδαμε τις συνέπειες ε, της, ε, του νέου νόμου. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του Σαββάτου είναι ότι η πλειοψηφία των δικαστών, 50 από τους 95, ψήφισαν υπέρ του καθηγητού Βότινες Βρούμπελ. Κατόπιν, ο, η δεύτερος προσηφίος, η καθηγήτρια Βαμανόφσκα, έλαβε 25 ψήφους. Μετά είχαμε τον καθηγητή Ντεμεντέντσκι που έλαβε 14 ψήφους. Ο πρώτος πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο ενδιάμεσος πρόεδρος, υπέβαλε 5 υποψηφίους στον πρόεδρο και ο πρόεδρος όπως ξέρουμε επέλεξε και όρισε ήδη την καθηγήτρια την κυρία Ταμανόφσκα. Προφανώς το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν είναι δεσμευτικό λοιπόν. Το τρίτο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να δείξω, είναι οι πειθαρχικέ διαδικασίες κατά δικαστών και εισαγγελέων. Θα ήθελα και πάλι να επανέλθω στον νόμο Φήμοτρο. Ε, δημιουργήθηκαν με αυτόν τον νόμο νέα πειθαρχικά παραπτώματα για τους δικαστές. Παραδείγματος χάρη είναι παράπτωμα οι δικαστές να εμπλέκονται σε δραστηριότητες οι οποίες είναι ασύμβατες με την αρχή της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας. Η νομοθεσία εισάγει την πειθαρχική ευθύνη των δικαστών όταν βγάζουν αποφάσεις οι οποίες είναι αντίθετες με τις προσδοκίες της πολιτικής εξουσίας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. 13 δικαστές ε, από ένα τόπικο δικαστήριο αντιμετωπίζουν πειθαρχική δίωξη επειδή έγραψαν μια επιστολή στον ΟΑΣΕ στην οποία ζητούσαν ο ΟΑΣΕ να παρακολουθήσει τις προεδρικές εκλογές και να στείλει παρατηρητές. Τώρα ο πειθαρχικός επίτροπος του δικαστηρίου Γκέτμπουργκ ερευνά τους δικαστές και ζητάει εξηγήσει. Την προηγούμενη εβδομάδα η ε, Επίτροπος ξεκίνησε προκατακτική διαδικασία καθώς θέλησε, ε, θεώρησε πως ε, η σύνταξη της επιστολής ήταν πειθαρχικό παράπτωμα, δηλαδή ήταν κάποιες ε, δραστηριότητες που είναι ασύμβατες με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνη. Ένα άλλο παράδειγμα αφορά μία εισαγγελέα, την Εύα Ζόζεκ. Είναι ανεξάρτητη εισαγγελέα από την Βαρσοβία, μέλος της Ένωσης Lex Super Omnia η οποία ξεκίνησε να έρευνα την οργάνωση της προεδρικής ε, εκλογής κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η έρευνα της αφαιρέθηκε αμέσως και απόφαση έβγαλε ε, μια άλλη εισαγγελέα απόφαση να σταματήσει η έρευνα. Μετά από τρεις ώρες εξέτασης της υπόθεσης και χωρίς να δει καν τους φακέλους. Τώρα, η Πειθαρχική Επίτροπο για του Εισαγγελεί έχει ξεκινήσει διαδικασία βάρος της ε, για την υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της. Το τέταρτο θέμα είναι τα προσωρινά μέτρα που ισχύουν από 8 Απριλίου και επηρεάζουν το καθεστώς των ε, δικαστών του πειθαρχικού τμήματος ε, του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Να σας πω μόνο το εξής. Μετά από την απόφαση αυτή, του δικαστηρίου στις 10 Απριλίου 2020 το πειθαρχικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου παρέπεμψε στο Συνταγματικό Δικαστήριο ένα νομικό ερώτημα για την δυνατότητα του ΔΕΚ να εφαρμόσει προσωρινά μέτρα για την λειτουργία της δικαιοσύνης ε, σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον τον Μάιο του 2020 ο πρώτος πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου ε, αποφάσισε επίσης πως ε, και οι πειθαρχικές υποθέσεις των δικαστών θα παραπέμπονται στην γραμματεία του Προέδρου όπου θα παραμένουν μέχρι να αποφασίσει το συνταγματικό δικαστήριο ή να απορριφθούν. Προφανώς το πειθαρχικό τμήμα αναμένει την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου. Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι όταν ενημερώθηκε για την απόφαση του ΔΕΚ ο πρόεδρος ε, Ντούντα όρισε τρεις ε, δικαστές στο πειθαρχικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Να αναφερθώ τώρα στην κατάσταση που αφορά την ελευθερία έκφραση στην Πολωνία. Ή όλοι ξέρουν πως η ελευθερία του συνέρχεστε έχει ανασταλεί ακόμα και δύο άτομα αν περπατούν στον δρόμο και κρατούν ένα πανό θεωρούνται παράνομη διαδήλωση. Υπάρχουν πολιτικοί λόγοι βεβαίως για την απαγόρευση διαδηλώσεων ενώ ταυτόχρονα η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία χαλαρώνουν τους περιορισμούς ε, για τους γάμους, ε, εκκλησίες κτλ. Η κατάσταση λοιπόν για το τραγούδι αυτό που αναφέρατε του Καζικ στο ραδιόφωνο μας δίνει ένα παράδειγμα για την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η κατάσταση, ο πόνος είναι καλύτερος από το δικό μου, αναφέρεται στην, ε, στο ότι είχαν κλείσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας όλα τα νεκροταφεία. Αλλά αυτό δεν αφορούσε τον επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος μπορούσε να πάει στον τάφο της μητέρας του, ενώ αυτό απαγορευόταν στους υπόλοιπους πολίτες. Το τραγούδι αυτό επελέγει από τους ακροατές της δημόσιας ραδιοφωνίας στα top 3 τραγούδια επειδή ασκεί κριτική ε, στο κυβερνών κόμμα. Για τον λόγο αυτό, την επόμενη μέρα ανακοίνωσε το, το πολωνικό ραδιοφωνό, έβγαλε το τραγούδι από τον λίστα και μετά την ακύρωσε. Ε, με συγχωρείτε κύριε Χεταρόβιτς, βεβαίως παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον όλα όσα λέτε, αλλά να έχετε κατά νου και τον χρόνο, γιατί έχουμε φτάσει στα όρια της τηλεοδιάσκεψης, έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο και θα δημιουργηθούν προβλήματα στο τέλος, γιατί υπάρχει άλλο ένα θέμα στη μερίσια διάταξη. Οπότε σας παρακαλώ να συντομεύετε. Λοιπόν, συμμερίζομαι και εγώ λοιπόν την ανησυχία που εξέφρασε ο εισηγητής ε, της ε, έκθεσης ε, όσον αφορά την κατάσταση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Πολωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. for having been sensitive <laughs> to the εμείς, εμείς σας ε, ευχαριστώ. Να σας ευχαριστούμε και συμπαθάτε που σας επισήμανα το ευαίσθητο, το λεπτό θέμα ε, του χρόνου αγορευσή. Και τώρα, πριν δώσουμε το λόγο στου συνοριστέ, θέλω και εγώ να λάβω το λόγο, γιατί είμαι ο εισηγητή. Όχι, όχι. Πρώτα-πρώτα να κάνουμε ένα γύρο τραπέζι και να ακούσουμε του ε, συντονιστέ. Πρώτα-πρώτα, κυρία Μετσόλα, για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τους προσκεκλημένους μας. Ε, ευχαριστούμε και εσένα, Χουάν Φερνάντο, που είσαι ο εισηγητής. Εμείς προβληματιζόμαστε βαθιά για την χώρα, για το το έχει αποκλίνει από τη δημοκρατική διακυβέρνηση για αυτόν τον νόμο φήμοτρο για τις επιπτώσεις στην δικαιοσύνη, τα σχετικά με το πειθαρχικό τμήμα, το ότι έχουν σταματήσει να απευθύνουν προδικαστικές ερωτήσεις, και η δίωξη όσων απευθύνθηκαν στο ΟΑΣΕ, στον ΟΑΣΕ σε σχέση με πρωτικές εκλογές, ε, όλα αυτά για τα όσα γίνονται εκεί. Εμείς παρακολουθούμε, ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ανασταλεί η λειτουργία αυτών των οργάνων που χρησιμοποιεί το καθεστώς και έχει επιβεβαιωθεί ότι ο κύριος Ντούντα τώρα, σήμερα, όρισε σε παραβίαση πάσης ε, παράδοσης και συνηθιών παρά τα όσα είπε η Ένωση Δικαστών, διόρισε τον πρόεδρο του το Τώρα βλέπουμε ένα κείμενο το οποίο έχουμε, θα γίνει συζήτηση μεταξύ πολιτικών δικαιωμάτων με αυτό το σχέδιο κειμένο ε, θα πρέπει να δούμε ε, την αρχή του κακού, όσα έγιναν με τις μεταρρυθμίσεις, όλα, όλα που δυναμίτησαν το κράτος δικαίου. Θεωρούμε ότι εκεί θα πρέπει να επικεντρωθεί η έκθεση, να δούμε πού έχει αρμοδιότητα η κοινοτική ένωση, πώς να είμαστε αποτελεσματικοί, αλλά κράτος δικαίου σημαίνει τήρηση κάποιων ε, προτύπων, κάποιων αξιών, κάποιων διατάξεων θα πρέπει να τηρηθούν δημοκρατικές διαδικασίες και έχουμε πει επανειλημμένα ότι δεν πρόκειται για κάποιες ιδέες αφηρημένες. Το θέμα είναι το πώς η Ευρώπη δεν θα ξαναπέσει στα ίδια λάθη τα ιστορικά. Ε, θέλω να ρωτήσω τον πρόεδρο Μάτος να μας εξηγήσει καλύτερα το τι ανταπόκριση υπήρξε στις παρατηρήσεις της Ένωσης Δικαστών, τι ανταπόκριση είχε από τις ε, πρώην αρχές. Επίσης θέλω να μας πει και η Κομισιόν ποιε ποιες είναι οι εξελίξεις όσον το διάλογο με την Πολωνία. Now, no further ado. Ευχαριστώ κύριε Μετσολά και χωρίς να καθυστερήσουμε να ακούσουμε τη φωνή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Να πάρει το λόγο η κυρία Σελβία Σπουρέκ, η συνάδελφό μα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και παρακολουθώ τη διαδικασία συστηματικών παραβιώσεων του κράτου δικαίου στην Πολωνία ω ε, μέλο ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και προηγουμένω ε, σε ό,τι αφορά την, ε, το δικαστικό, το δικαστήριο το μονοπόλιο σε ό,τι αφορά την ε, διορισμό δικαστηρίων, ε, η δυσφήμιση των δικαστών, αυτός ο πρόσφατος νόμος φήμοτρο, αλλά και ο περιορισμός του ε, χώρου του πολιτικού χώρου, η παραβίαση της συνθήκης της Κωνσταντινούπολης, ο περιορισμός των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ, είναι πραγματικά ο κατάλογος ατέρμονος. Και όλα αυτά δυσχρένονται από το COVID και η πολωνική και η ουγγρική κυβέρνηση απομακρύνονται όλο και πιο πολύ από τις δημοκρατικές αρχές και δεν έχουν αντιμετωπίσει καμία, αμ, κανένα αντίπεινο. Έχει έρθει λοιπόν η στιγμή να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν φτάνει να παρακολουθεί την κατάσταση. Θα πρέπει να απαιτήσει συμμορφώση και να υπάρξει αιρεσιμότητα με τους ευρωπαϊκούς πόρους. Πώς σχολιάζετε λοιπόν αυτά τα μέτρα, ποια θα μπορούσε να είναι μια αποτελεσματική λύση για την κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα να περάσουμε στον συντονιστή από το Ρενιού. Η κυρία Σοφή Ιντφέλτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και να σας ευχαριστήσω και ως εισηγητή για το θέμα αυτό. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το θέμα αυτό το συζητάμε τέσσερα χρόνια πλέον, αν δεν κάνω λάθο. Ίσως και παραπάνω. Και φαίνεται ότι η πολωνική κυβέρνηση δεν κόπτεται, για να το πω ευγενικά, για την ένωμη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ένα συμπέραγμα εξαγάγω μόνο. Αν δεν αποδεχόμαστε πλέον την αρχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση των συνθήκων, δεν θέλετε να είστε μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον ουσιαστικά. Δεν μπορείτε να ενεργείτε εκτός του νομικού πλαισίου και να είστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλα τα πλεονεκτήματα συμπεριλαμβανομένης και της ε, παροχής πόρων. Και αυτό λοιπόν φέρνει στα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα το κατά πόσο θα μπορούσε να επιθέλθει μια ρήτρα αιρεσιμότητα για το κράτο δικαίου στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και νομίζω ότι σύντομα θα κληθούμε να ψηφίσουμε το ευρωπαϊκό πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε η ρήτρα αιρεσιμότητα να μπει ω τμήμα του ΠΔΠ. Ο κύριος Ντεμάτος ζήτησε ένα σχέδιο Μάρσαλ για το κράτος δικαίου. Θα ήθελα να υποστηρίξω την έκκληση αυτή. Και την προηγούμενη εβδομάδα η ομάδα Renew ενέκρινε μία έκκληση για να σχέδιο δράσης ε, κρίσης για το κράτος δικαίου. Γιατί βρισκόμαστε σε κρίση, όχι μόνο με την Πολωνία και την Ουγγαρία, υπάρχουν και άλλα θέματα. Αν υπάρχει λοιπόν μια κρίση, χρειάζεται και ένα σχέδιο αντιμετώπιση τη κρίση. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει ένα ε, γενικότερο σχέδιο και τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει και άλλα μέσα στην διάθεσή της στη διαδικασία επιπαραβάση. Καταλαβαίνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει κάποια μέτρα ήδη, αλλά είναι υπερβολικά αργά και περιορισμένα και υπάρχουν και άλλες παραβιάσεις. Δεν έχει να κάνει μόνο με την κατάργηση της ανεξαρτησίας των δικαστών στην Πολωνία. Είναι πλέον η Πολωνία ε, μια κατόνομα μόνο δημοκρατία αλλά και τα δικαιώματα των γυναικών, το δικαίωμα άμβλωσης και καθορισμού της ε, τύχης του σώματός τους και της ζωής τους. Απόπειρε για την χειραγώγηση της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου, περιορισμού, περιορισμός της ελευθερίας έκφρασης των ΜΚΟ, ακαδημαϊκής ελευθερίας, είναι πραγματικά κατάλογος πολύ μεγάλος και νομίζω ότι είναι σαφές πλέον από πλευρά του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι το άρθρο 2 αποτελεί δικαστική ε, νομική βάση, το οποίο θα μπορούσε και θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναλάβει δράση. Ευχαριστώ με την κυρία Εντφέλντ. Σας ευχαριστώ κυρία Εντφέλντ. Ε, Τώρα θα ακούσουμε τον συνάδελφο, τον κύριο Νίκολας Μπέι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη προσοχή άκουσα τους ε, προελίσσαντες ε, και τις επικρίσεις που διατύπωσαν για το πώς τροποποίησε, πώς άλλαξε την οργάνωση της ε, δικαιοσύνη. Εδώ πριν από δύο χρόνια πήγατε στην Βαρσονία, κάνατε την αποστολή και υπήρχαν πάρα πολλοί αντίπαλοι του ΠΙΣ ε, με τους οποίους είχατε μιλήσει και επίση υπήρχε φόβος, φόβος ε, σε σχέση με όλες αυτές τις ε, ενέργειες αυτούς και, και σήμερα ακούσαμε δύο που επικρίνουν και όμως δεν έχουμε απάντηση επίσημη όπως και τότε και οπότε όλα θα το κάνει η Πολωνία. Μπορεί να φτιάχονται ε, κριτική αλλά και στη Γαλλία ε, έτσι ε, γίνεται ε, έτσι ορίζονται οι ανώτατοι δικαστές από τον πρώτο Δημοκρατίας, οπότε επίσης και στην Ιταλία αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε δύο δικαστές που ε, είχαν ε, κάνει κάποιες παρασπονδίες όσον αφορά το μεταναστευτικό, αλλά ήταν δύσκολο να βρεθεί ένας τρόπος να καταδικαστούν αυτοί. Και οπότε ε, τελικά οι επικρίσεις παίζουν ρόλο στις εκλογές. Είπατε κυρία Ινετφέλτ για τους LGBTI, για τους ΛΟΑΔΚΙ, αλλά όχι, όχι, το θέμα δεν είναι η κάθε μια κατηγορία χωριστή. Οι Πολωνοί κάνανε εκλογές, ψηφίσανε, ενέκριναν τις ε, αλλαγές στη δικαιοσύνη. Βεβαίως και θα ληφθούν υπόψη επικρίσεις, αλλά στη δημοκρατία ε, τον τελευταίο λόγο τον έχει ο λαός. Δεν θα πρέπει στα θεσμικά όργανα να προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε ε, και να βάλουμε τους εαυτούς μας στη, στη θέση του λαού. Για το άρθρο 7, ξέρετε, δεν υπάρχει συνένεση. Δεν πρέπει να προχωρήσουμε προς τα εκεί. Θα πρέπει να τηρηθούν οι συνθήκες και από το Κοινοβουλίο. Αν δεν υπάρχει η συνένεση, τι να κάνουμε. Καλά, μπορείτε να επικρίνετε την κυβέρνηση εκείνης της χώρας, αλλά δεν μπορεί να κάθεται στο εδόλιο κάποια χώρα που έχει θέση στην Ευρώπη σε σχέση με τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη στο μέλλον. Merci, Monsieur Bay. Ε, have been reported that. Ε, Σας ευχαριστώ. Μου λένε εδώ ότι υπάρχει ένα τηλεοπτικό συνεργείο από την Πόζακ, έναν πολωνικό ε, τηλεοπτικό σταθμό που παρακολουθεί τη συζήτησή μας και ε, καταγράφει τα όσα δείχνει η οθόνη. Να το έχετε λοιπόν κατά νου. Μεταδίδεται λοιπόν η συνεδρίασή μας ζωντανά. Περνάμε τώρα στους πράσινους. Η κυρία Στρίκ, φαντάζομαι. Με ακούτε, έχετε τον λόγο. Όχι, η κυρία Ράντκε θα είναι. Έτσι τα είχαμε πει. Τα είχαμε πει στη γραμματεία. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Να, να. Να με συγχωρείτε. Εδώ μου είχαν σημειώσει στρικα. Δεν ξέρω, η κυρία Ράντ και με ακούει. Εδώ είμαι, ελπίζω να με ακούτε. Να κάνω το εξή σχόλιο. Ε, συνεχώς ακούμε ότι δεν δίνεται χώρος στα άτομα τα οποία εκφράζουν τις απόψεις πολωνικής κυβέρνησης. Ε, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί έχουν κληθεί πολλές φορές, αλλά δεν απαντούν τις ερωτήσεις ε, και τις αποφεύγουν. Και αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζουμε. Τώρα προς ε, τους ομιλητές ε, της σημερινής συνεδρίασης σας ευχαριστώ και θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Ίσως λοιπόν εδώ πέρα έχουμε μια αυθύνουσα πορεία. Αν συνεχιστεί αυτό, ε, θεωρείτε ότι μπορούμε να μιλάμε για ένα κύμα αυταρχισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζητήματα κράτους δικαίου και φιλελεύθερης ε, δημοκρατίας, κάτι το οποίο ανησυχεί πάρα πολλούς. Και προς ε, τον συνάδελφο που αναφέρθηκε ε, για την ε, δημοσιονομική αιρεσιμότητα θεωρείτε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο για να ελεγχθεί η κατάσταση. Και βεβαίως όσον αφορά την ατμόσφαιρα μεταξύ των πολλών δικαστών γνωρίζουμε ότι είναι σοβαρές οι πιέσεις να δούμε τι μπορεί να γίνει τέλος προς τον κύριο εισηγητή θα ήθελα να επαναλάβω και πάλι το θέμα της κατάστασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, οι ζώνες ε, ελεύθερες από ΛΟΑΤΚΙ. Θεωρώ πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ζητήσει διαδικασία επί παραβάση ε, με βάση την νομοθεσία περί διακριτικής ε, μεταχείρισης. Δεν έχουμε μια σχετική οδηγία, αλλά υπάρχει νομοθεσία για διακριτική μεταχείριση πύχη στην αγορά εργασία και θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει σχετικέ διαδικασίες γιατί οι Πολωνοί πολίτε και οι ΛΟΑΤΚΙ τέτοιοι πρέπει να προστατεύονται από την ε, νομοθεσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ για το ECR τώρα. Ο κύριος Γιάκε, έχετε τον λόγο, εάν με ακούτε. Πιέσατε το κομβίον, παρακαλώ. Τώρα, με ακούτε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους προλαλήσατες. Βεβαίως οφείλω να διαμαρτυρηθώ για την ε, παρουσίαση αυτής της έκθεσης. Βλέπω εδώ πέρα παραδείγματος χάρη πως ε, Το Ιουστίτσια τώρα μίλησε για ακροδεξίες ενώσεις, δεν ξέρω τι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι αντιεπαγγελματικό και από την πλευρά της έκθεσης νομίζω ε, το να παρουσιάζεται η κυβέρνηση ως ε, κάποια η οποία ε, παραβιάζει το Σύνταγμα. Πολύ απλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το Συμβούλιο Δικαιοσύνης δεν είναι δικαστήριο το ίδιο. Το ένα είναι αυτό. Το γνωρίζετε αυτό άλλωστε και με κάθε σεβασμό για τον ε, πρόεδρο. Μα εκλέγεται όπως εκλέγεται και στην Ισπανία άλλωστε. Αυτό το κάνει το κοινοβούλιο. Η διαφορά είναι μάλιστα ότι είναι με απλή πλειοψηφία στην Ισπανία ενώ απαιτούνται τρία πέμπτα στην ε, Πολωνία. Το δε κόμμα ε, δεν υπερψήφισε. Οπότε πώς είναι δυνατόν να είναι εντάξει στην Ισπανία αλλά όχι στην Πολωνία. Ε, δηλαδή εξηγήστε το αυτό. Και επίση ε, έχουμε και το συνταγματικό δικαστήριο στο άρθρο 15, μετά έχουμε το άρθρο 21, ε, το οποίο ακριβώς αντιφάσκει με την τελευταία απόφαση του ΔΕΚ. Ε, μα πώς γίνεται αυτό είτε δεχόμαστε και αναγνωρίζουμε το ΔΕΚ, είτε όχι. Το συνταγματικό δικαστήριο, με συγχωρείτε, είτε όχι. Γιατί το συνταγματικό δικαστήριο συμφωνεί με την πολωνική κυβέρνηση. Και μετά στο σημείο 16 λέτε πως ήταν απόφαση του Προέδρου ε, η εκλογή του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Μα αυτό, ε, το γράφει το Σύνταγμα από το 1990. Το άλλο επίσης που πρέπει να αποφασίσετε είναι αν ε, επιτρέπεται να τοποθετούνται πολιτικά οι δικαστές. Ε, το πολωνικό σύνταγμα το απαγορεύει ας πούμε αυτό. ένα κείμενο του 1997. Τώρα, ε, εκτρώσεις, ε, σεξουαλική αγωγή, ούτε αυτό ισχύει. Πρέπει να τηρήσουμε την πολωνική νομοθεσία. Αυτό δεν είναι στήριξη στην κυβέρνηση. Αν υπάρχει μια πρωτοβουλία πολιτών τους χάρη, ναι, η οποία αφορά την Ισπανία, την Αφρική, Κοιτάξτε, ή αν υπάρχει μια συμφωνία εμπορική, πρέπει να την τηρήσουμε. Δεν σημαίνει αυτό ότι συμφωνούμε ή όχι. Όσον αφορά τώρα τις εκτρώσεις, και με στην κοιλιά της μητέρας ε, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ανθρώπινα δικαιώματα. Yes, yes, yes, now. Μάλιστα. Διακόπτη πρόεδρος. Now we move to... Μάλιστα, λοιπόν, λέει ο πρόεδρος. Να περάσουμε τώρα στον επόμενο συντονιστή. Από την ΚΟΕ. Η Κορνίλια Έρνης, αν δεν κάνω λάθος. Mrs. Ernst, may I kindly ask you to... Κυρία Ernst, το πλήκτρο speak, αν θέλετε. Mrs. Ernst, if there is any problem, Κυρία Ένστε, αν υπάρχει πρόβλημα, προτείνω το εξή. Έχω άλλο ένα μέλος, θέλει να πάρει το λόγο για ένα λεπτό μόνο. Αν θέλετε να πάρει πρώτα το λόγο και μετά να ακούσουμε και εσάς, πρώτο παρά το λόγο εγώ ως εισηγητής. Ο συνάδελφος Πολ Ραντζέλ θέλει να πάρει το λόγο για ένα λεπτό. Αν καταλάβω σωστά. Αν έχετε λοιπόν σύνδεση, μπορείτε να πάρετε το λόγο. Nope It doesn't seem to be the case. Δεν έχει μάλλον σύνδεση. Η κυρία Ένστ από την ΚΟΕ είναι έτοιμη να πάρει το λόγο. Μας ακούτε. Okay, then please Μάλιστα. Να πάρω εγώ το λόγο ω συζητητή. Για να σας παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία της ε, έκθεσης αυτής, η οποία είναι έτοιμη να προσαρμοστεί ανάλογα και με τις τροπολογίες σας ε, με τη σύναψη συμβιβαστικών ε, λύσεων. Η διάμεση λοιπόν αυτή η έκθεση, το σχέδιο έκθεσης. Ακολούθησε την διαδικασία του άρθρου 7 παραγραφός 1 σε σχέση με την Πολωνία. Προσπάθησα να αναφέρω διάφορες ε, διαστάσεις των εξελίξεων που δυστυχώς επηρέασαν αρνητικά τα θεμελιώδη δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τα δημοκρατικά δικαιώματα στην Πολωνία. Αυτό όχι μόνο τους τελευταίους μήνες, αλλά πλέον πάνε χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με την κατάσταση αυτή, δυστυχώς. Έχουμε και τις ε, καταστάσεις τις οποίες επισημαίνουν και ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις, ε, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Επιτροπή στο ECE. Είναι με τα Έθνη, η ΟΝΤΙΡ, Έχουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τα διεθνή δικαστήρια και άλλα δικαστήρια που έχουν ε, καταδικάσει τις καταστάσεις αυτές. Ε. Έχουμε επίσης ε, κάνει διαβουλεύσεις με τις πολωνικές αρχές. Όταν η Μπέατα ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, άκουσα με προσοχή και συμμετείχα στη συζήτηση αυτή. Το ίδιο και το Ματέος Μουραβιέσκη, τον επόμενο Πρωθυπουργό και με τον κύριο Τζιόπρο, τον ε, Υπουργό Δικαιοσύνη. Ακούσαμε και τα δικά του λόγια. Κύριε Καλέτα, προσφάτως και φυσικά εκπροσώπους της πολιτικής κυβέρνησης που είχαν πάσα ευκαιρία, κάθε ευκαιρία να διαλευκάνουν όλα τα ζητήματα τα οποία είχαμε εκφράσει ως ανησυχίες από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και παρά όλα αυτά κάποιες ερωτήσεις οι οποίες θέσαμε δεν απαντήθηκαν ποτέ. Εγώ, για παράδειγμα, θυμάμαι ότι για να κλειτώσουμε χρόνο είχα ε, ζητήσει να μου απαντήσουν μόνο δύο συγκεκριμένα στοιχεία. Προς τον κύριο, α, ε, τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, όταν εμφανίστηκαν στην Επιτροπή α, ε, ΛΥΜΠΕ και ούτε μία από αυτές τις δύο ερωτήσεις τις οποίες έθεσα εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής δεν απαντήθηκαν. Δεν απάντησαν σε καμία από τις δύο ερωτήσεις. Για τη συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε ό,τι αφορά το πτωρχικό σώμα και την απόφαση που έλαβε η πολωνική κυβέρνηση να απαντήσει στη διαδικασία επιπαραβάση και στη σχετική δικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Άρα ακούσαμε τα θεσμικά όργανα, τους ε, δικαστές, ε, τους νομικούς, την κοινωνία των πολιτών, τους δημοσιογράφους και σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, σε ό,τι αφορά και την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, η κατάσταση στην Πολωνία δεν βελτιώνεται. Αντιθέτως, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες Το 2015 ξεκίνησε το θέμα αυτό για τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Δικαστικού Σώματος σε ό,τι αφορά το... τις διαδικασίες εισαγγελής ε, και το θέμα των πειθαρχικών μέτρων κατά των δικαστών που εξέφρασαν τη γνώμη τους κατά των μέτρων αυτών. Και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι κανένα από τα θέματα αυτά δεν μπορεί να ειδωθεί ξεχωριστά. Δεν μπορεί να το εξετάσουμε μεμονωμένο. Γιατί αποτελεί τμήμα μιας στρατηγικής, η οποία εκτελήσεται σε ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο τα τελευταία χρόνια. Έχουν ληφθεί λοιπόν τέτοιες αποφάσεις. Δεν είναι θέμα λοιπόν μόνο της μία ή της άλλης απόφασης εκείνου ή του άλλου μέτρου ή της συμβατότητας ενός και μόνο μέτρου με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το θέμα είναι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν λάβει η χώρα αυτό το χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν διακρίνουμε ε, ένα pattern, διακρίνουμε μια σταθερή συμπεριφορά θεσμικών αλλαγών οι οποίες όλες αποσκοπούν προς την ίδια κατεύθυνση. Έναν στόχο. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Και άρα λοιπόν έχουμε τις εξής συνέπειες, οι οποίες επίσης διευκρινίζονται στο άρθρο 7 της συνθήκης για το δικαστικό σώμα. Συστημική λοιπόν και κατάφορη παραβίαση του κράτους δικαίου σε ό,τι αφορά την επιρροή με κρίσιμο τρόπο στις εργασίες του δικαστικού σώματος. Και έτσι λοιπόν τύφεται ένα αμφιβόλο η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος. Αυτή η θεσμική διαφορά λοιπόν στην Ευρωπαϊκή, Επίτρο... στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί στις προνοικές αρχές ε, αρέσει να κάνουν ε, σύγκριση και με άλλε κυβερνήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, αυτή η γενική τάση δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο κράτο μέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλε οι χώρε ε, έχουν ε, αδύναμα σημεία, στοιχεία τα οποία χρήζουν κριτική ενδεχομένω. Αλλά πρόκειται για μη συστηματική απόπειρα ελέγχου ολικού ελέγχου του δικαστικού σώματος και είμαι πεπισμένος ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 η νομοθεσία που έχει περάσει σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι για παράδειγμα στο θέμα των αμβλώσεων, των αρμοδιοτήτων του Προέδρου κτλ. Και στον ένα αυτό πλαίσιο οι πολίτες δεν ε, λειτουργούν πλέον σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι συμβατό με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι άλλο που είναι πολύ σοβαρό για την οργάνωση των προεδρικών εκλογών και σε ό,τι αφορά το πλαίσιο της πανδημίας. Εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση ανεξάρτητων αμερόληπτων εκλογών την Πολωνία ότι αυτό δεν ήταν δυνατόν να λάβει χώρα. Σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, η προτινόμενη νομοθεσία για, την, αμα, για τις αμβλώσεις ουσιαστικά ισοδυναμεί με απαγόρευση πλήρη της των αμβλώσεων. Σε ό,τι αφορά επίσης το επίπεδο προστασίας των μειονοτήτων, τα δικαιώματα των ε, γυναικών, τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΑ, τα κράτη-μέλη έχουν και ηθική αλλά και νομική υποχρέωση να προστατεύσουν την ηθική και σωματική ακυρεότητα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανόμενα και των Πολωνών. Το δικαίωμα στα δική δίκη, ελεύθερη του συνέρχεστε, ελεύθερη του τύπου, και το τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι η πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Γι' αυτό θέλουμε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής αυτής για να συμπεριληφθεί και το άρθρο 7 παράγραφος 1 για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλούμε προφανώς την πολωνική κυβέρνηση με όλο τον δέοντα σεβασμό να συμμορφωθεί με όλες τις διατάξεις που έχουν να κάνουν με το, καθώς δικαίωτο το τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις δημοκρατικέ ελευθερίες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ή χρειάζεται λοιπόν να υλοποιηθούν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να υπάρξει σεβασμός και του ιδιωτικού δικαίου, το οποίο επίσης διακυβεύεται από τον επωνομαζόμενο νομοφήμοτρο, προκειμένου τελικά να υπόκεινται κυρώσεις οι δικαστές οι οποίοι α, αμφισβητούν τα νομοσχέδια. Αυτό αποτελεί λοιπόν σημαντική αξία και σημαντική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλούμε λοιπόν το Συμβούλιο να δράσει στα πλαίσια του άρθρου 7 παραγράφου 1. Σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, αντιμετωπίζοντας τις συγκεκριμένες ε, συστάσεις. Καλούμε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα μέσα που έχει στη διάθεσή του και να ξεκινήσει διαδικασίε ε, επί παραβάση, χρησιμοποιώντα και τις δημοσιονομικές δυνατότητες που έχει, όπως έχουν συζητηθεί τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ε, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει όπως ε, δει. Με όλο το σεβασμό προς την κυβέρνηση της ε, Πολωνίας έχει έρθει η στιγμή να δράσουν και να μην επιδείξουν ε, ασέβεια προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, μας, ε, τους εκπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων των Πολωνών πολιτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Now τώρα να δώσουμε το λόγο ξανά στους ε, προσκεκλημένους μας ε, Μάτος Ετνάροβιτς για να μας ε, απαντήσουν, να τοποθετηθούν σε αυτά τα οποία άκουσαν. Έχετε ξανά το λόγο. Mr. Arvanitis, may I kindly ask you to... Κύριε Αρβανίτη, πρέπει να πατήσετε το κουμπί που λέει speak. Κύριε Αρβανίτη, σας ευχαριστούμε. Έγινε ένα μικρό λάθος. Ε, χαιρετώ όλους τους συναδέλφους και τον ε, Πρόεδρο φυσικά. Κοιτάξτε κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, το σημερινό θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και η εισήγηση, η προσωρινή έκθεση αναγνωρίζουν το ιστορικό βάρος από, την συγκεκριμένη, από μια συγκεκριμένη άποψη, τη θεσμική, το θέμα είναι πιο δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και από αυτή του Brexit. Κατά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είχε τεθεί θέμα δοκιμασία των καταστατικών αρκών και πυλώνων τη ΕΕ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζητούμενο, όχι για πρώτη φορά, το θέμα τη Πολωνία, δηλαδή, ε, ωστόσο, όντω αφορά το άρθρο 2 τη ισχύουσα ενοποιημένη συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι αξίε τη αξιοπρέπεια της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Τις αρχές δηλαδή που συνθέτουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Συμφωνώ μάλιστα ανεπιφύλακτα με την αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής της 17ης 12 του 2017 πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει και άλλους κινδύνους παραβιάσεων της δημοκρατίας και, το, και του κράτους δικαίου. Καταλαβαίνω μια νοστόρα διστακτικότητα εξαιτία του λεγόμενου διλήμματος της Κοπενχάγης, αλλά τα περιθώρια πλέον τέλειωσαν. Δεν υπάρχουν δικαιολογίε αφού είναι λογικά αυτονόητο ότι οι θεμελιακοί όροι εισδοχή ενός μέλους αποτελούν και τους λόγους παραμονή του. Στην Πολωνία, η συνταγματική αναθεώρηση με μη προβλεπόμενο τρόπο, ο κυβερνητικό έλεγχος της δικαιοσύνη, οι προσβολές δικαιωμάτων έκφρασης και συνένωση, οι στευλή όρη οργάνωση εκλογών, όλα αυτά συνιστούν όχι εφάπαξ, αλλά συστημικά πλήγματα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, τα οποία αντανακλούν ευθέω στα θεσμικά κείμενα τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα κράτη-μέλη. Εξάλλου γνωρίζω τι εκτάκτε συνθήκε που συνδέονται με τον COVID, αλλά αυτέ καθόλου δεν συνδέονται με τα συστημικά θέματα λειτουργία, τη νομοθετική και δικαστική λειτουργία, ώστε να υποχρεώνουν σε, αφορ... σε αφόρητε κάμψει του. Κλείνοντα, είναι σημαντικό το γεγονός ότι η προσωρινή έκθεση προχωρεί στο άρθρο 1 σε εξειδίκευση των φυγόμενων αρχών, λειτουργία νομοθετικών και εκλογικών αρχών, ανεξαρτησία δικαιοσύνης, θέματα κράτους δικαίου, ώστε να είναι δυνατό να στηριχθούν στη διάγνωση συγκεκριμένων παραβιάσεων αφενός, η κίνηση διαδικασίας και μηχανισμού ελέγχου, κατά το άρθρο 7, παράγραφος 1 της ΕΕ και αφιτέρου η λήψη σχετικών μέτρων που αφορούν το προπολογισμό τη Ένωση. Μία απάντηση προ του Πολωνού φίλου μα. Μην αναφέρεστε όταν, απαξιωτικά όταν αναφέρεστε στου Ευρωβουλευτέ και στο Ευρωκοινοβούλιο και μην αναφέρεστε συνέχεια στο πρόσφατο παρελθόν σα που είχατε αυτό το λεγόμενο κομμουνιστικό καθεστώ καρικατούρα δημοκρατία. Όλε μα οι χώρε έχουν τα βάσανά του και τι πολύ άσχημε ε, ιστορικέ στιγμές. Εμεί είχαμε Χούντα, οι Ισπανοί είχαν το Φράγκο, οι Ιταλοί είχαν το Μουσολίνι. Προχωράμε όμω. Αυτό δεν μπορεί να γίνει καραμέλα για δημοκρατίε τύπου Ρωσία, Πούτιν ή άλλου τύπου που είναι έξω από τα δικά μα πλαίσια. Συμφωνώ και είμαι θετικό στην ε, κεντρική εισήγηση του Προέδρου μα. Σας ευχαριστώ. χαθεί η εικόνα. Ο πρόεδρος. Κύριε Αρβανίτη, σας ευχαριστούμε. Και ο κύριος Ρανζέλ νομίζω θέλει το λόγο. Παρακαλώ μέχρι ένα λεπτό, κύριε συνάδελφε. Κύριος Ρανζέλ. Δεν ακούει το κύριο Ρανζέλ. Μ' ακούτε, μ' ακούτε. Α, ωραία. Μια χαρά. Μ' ακούτε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλώς, ευχαριστώ. Σας ακούμε, σας ακούμε. Προχωρήστε. Λέει ο πρόεδρος. Δεν εκπλήσωμε που ήρθε εδώ ο κύριος ε, Μάτος, τον ξέρω πολύ καιρό και ανέκαθεν έδινε μάχη για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και για την υπεροχή του κράτους δικαίου. Οπότε καλωσόρισε, καλωσόρισε ο, ο κύριος ε, Μάτος και πάλι. Επίσης πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ με όλα όσα είπε η κυρία Μετσόλα. Και πρέπει να προσθέσω ότι αξίζει να προσέξουμε όχι μόνο τα θέματα της δικαιοσύνης, αλλά τα θέματα του κράτους δικαίου, την δημοκρατία στην Πολωνία. Γιατί τα θέματα αυτά είναι αλληλοσυνδεόμενα. Έχουμε αυτές τις πρόσφατες απόπειρες διενέργειας εκλογών σε πολύ περίεργες συνθήκες, στην επιστολική ψήφα. Αυτά είναι απαράδεκτα. Αυτή η επίθεση στην εξαρτησία της δικαιοσύνης είναι πάρα πολύ σημαντική για την υπεροχή του κράτους δικαίου στην Πολωνία. και θα πρέπει ευρύτερα να το δούμε το θέμα. Και πέστε μας εσείς κύριε Γκρέζα Μάτος, γίνεται στο μέλλον να έχουμε κάτι σαν μόνιμο μεχανισμό αξιολόγησης του αν ισχύει το κράτος του δικαίου της ε, ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε με τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι κάποιες χώρες θεωρούν ότι υφίστανται διώξεις. Έτσι λένε κάποιες κυβερνήσεις. Να υπάρξει ένας μηχανισμός που να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Έτσι. Πιο εύκολα θα παρακάμψουμε αυτές τις ε, ενστάσεις. Πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα να υπάρξει ένας τέτοιος μηχανισμός για όλους, για παρακολούθηση, για αξιολόγηση της κατάστασης του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας σε όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα και τώρα, οι προσκεκλημένοι μας. Σύντομες απαντήσεις σε όσα ακούσατε. Αλλά και σε σχέση με τα όσα είπα για την έκθεσή μου Και στη συνέχεια ως πρόεδρος και ως εισηγητής πρόκειται να εξαγάγω μετά κάποια συμπεράσματα. Πρώτα πρώτα η πρόεδρε Γκρέζα Μάτος, πρόεδρε της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών. Ξανά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα προσπαθήσω να απαντήσω στι ερωτήσει τι οποίε ε, άκουσα και να κάνω και κάποια σχόλια γενικά. Κυρία Μέτσολα, με ρωτήσατε σε σχέση με τις παρατηρήσεις ε, που έκανε η πολωνική κυβέρνηση σε σχέση με τις δηλώσεις μας. Η... Ξεκινήσαμε το 2015 σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του α, δικαστηρίου και προσπαθήσαμε να αναφερθούμε και στις, ε, να στραφούμε και προς τις πολωνικές αρχές για να λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις μας. Δυστυχώς δεν λάβαμε απάντηση από το 2015 μέχρι και σήμερα. Ε, κάνουμε εκτεταμένο διάλογο, αλλά προφανώ για το διάλογο χρειάζονται δύο μέρη. Και δυστυχώ ω σήμερα δεν έχουμε λάβει ουσιαστικέ απαντήσει από τι πολωνικέ αρχέ. Άρα έχουμε τι ίδιε εμπειρίε να αναφέρουμε, όπω και ο πρόεδρο τη Επιτροπή. Δεν έγινε ουσιαστικά διάλογο, μόνο αναβολέ. Επί αναβολών σε ό,τι αφορά τι απαντήσει, τι ερωτήσει που είχαμε θέσει και τελικά μας έφερναν διαρκώς πρώτο τελεσμένου. Και σε τελική ανάλυση έκαναν τις μεταρρυθμίσεις τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούμε να αντιδράσουμε. Δεύτερη ερώτηση από πλευράς της κυρίας Ρενκή. Και αυτή πολύ σημαντική για τις άλλες χώρες. Γιατί σήμερα αντιμετωπίζουμε το εξή πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η Πολωνία, είναι και η Ουγγαρία από ό,τι ξέρετε που έχει αυτοκρατικό, ε, αυταρχικό καθεστώς. Και αντιμετωπίζουμε λοιπόν πολλά τέτοια προβλήματα σε πολλές χώρες σε κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Αυτό το φαινόμενο copy-paste, όπως σας είπα, 60% των 44 χωρών σε ερωτηματολόγιο που αποστήλαμε στα μέλη μας, δήλωσαν τα τελευταία πέντε χρόνια έχει χειροτερεύσει το θέμα της δικαστικής ανεξαρτησίας. Δεν ξέρουμε τι είδου καθεστώτα θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Αλλά προφανώς όλων τα μάτια είναι στραμμένα στο τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Πολωνία και την Ουγγαρία. Αν δεν καταφέρουμε να προασπιστούμε την κοινότητα των καλών αυτών πολιτών, να στραφούμε λοιπόν και να προασπιστούμε ε, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, θα είναι και άλλες χώρες που θα ακολουθήσουν και ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε ένα σοβαρό πρόβλημα στο μέλλον με την δημοκρατία. Και αυτό είναι μια σημαντική πτυχή, την οποία και την υπογραμμίζω. Προφανώς η δημοκρατία και η νομιμότητα της δημοκρατίας κατοχυρώνεται με τις εκλογές. Και αυτό δεν το σχολιάσαμε. Όλοι όμως γνωρίζουν και μάλιστα το γράφουν και όλα τα σχετικά κείμενα ότι το θέμα δεν είναι μόνο οι εκλογές. Έχουμε το θέμα το, της διάκρισης των εξουσιών, το θέμα της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν αυτά, αυτοί οι πυλώνες, αν δεν είναι κατοχυρώνεται ο δεύτερος πυλώνας αυτός, δεν θα υπάρχει στη τελική ανάλυση δημοκρατία. Όταν ξεκινήσει αυτή ιδέα της δημοκρατίας. Η τυραννία της ε, πλειοψηφίας αποτελεί πάντα μια απειλή για τη δημοκρατία και η προάσπιση των ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου, του πολίτη, είναι κρίσιμη σημασία για να μπορέσει μια χώρα να αυτό αποκαλείται δημοκρατία. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω γρήγορα είναι αυτή η επιλεκτική χρήση, την οποία βλέπουμε συχνά Δίνονται δηλαδή κάποια ε, περιστασιακά παραδείγματα για άλλα θεσμικά όργανα, για άλλες χώρες και μας κατηγορούν ότι και άλλοι το ίδιο κάνουν. Τα τελευταία χρόνια έχω συνομιλήσει με εκατοντάδες δικαστές στην Πολωνία και είχα συναντήσεις με πολλούς εκπροσώπους από διεθνείς οργανώσεις, από εθνικές οργανώσεις στη χώρα και γνωρίζω πώς λειτουργεί το Δικαστικό Συμβούλιο στην Πολωνία. Ξέρω για παράδειγμα ότι ο Υπουργό Δικαιοσύνη πρόσφατα αντικατέστησε τον πρόεδρο του δικαστικού, της Δικαστικής Επιτροπής και προσπαθούν να τους ευρεάσουν με τρόπο ώστε να, καταργηθεί ουσιαστικά η αμεροληψία και η ανεξαρτησία τους και σε, σε μερισμένε περιπτώσεις και περιστάσεις. Αυτές οι ιεραρχικές δομές οι οποίες προσπαθούν να καθιερώσουν στην ε, Πολωνία ε, είναι πραγματικά ανησυχητικέ. Είναι πολύ διαφορετικέ ε, από ό,τι στην Ισπανία, για παράδειγμα. Ξέρω ότι πέρα από το σύστημα διορισμού του Δικαστικού Συμβουλίου, το Μαλακών Δικαστικού Συμβουλίου, στην Ισπανία είναι ουσιαστική η ανεξαρτησία των δικαστών. Γιατί πρόκειται για επαγγελματίε δικάστε, οι οποίοι ακόμα και όταν φεύγουν από το Συμβούλιο, λειτουργούν ως ανεξάρτητοι δικαστές και θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι δίκαιο το να συγκρίνουμε την Πολωνία με την Ισπανία και τέλος προς τον Παουλ Ρανζέλ, αγαπητό μου φίλο εδώ και χρόνια. Χαίρομαι πάντα που σας βλέπω και που παρακολουθώ και το έργο σας για το κρατός δικαίου. Έχω να σας πω το εξή. Είμαι πρόθυμος, πρόθυμότατος και είναι και θετική θεωρώ εξέλιξη να υπάρχει ένα μόνιμο μηχανισμό για την παρακολούθηση του κράτου δικαίου. Ε, είχαμε και μια συνάντηση με την Επίτροπο ε, Γιούρεβα και τον Επίτροπο Ρέιντερ για το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο και θα πρέπει να υλοποιηθεί γρήγορα, ταχύτατα. Γιατί θα μπορούσε να είναι πολύ ωφέλιμο. Ωστόσο, Ωστόσο και με αυτό θα κλείσω. Επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχει πραγματικά κατεπήγον χαρακτήρα στο θέμα αυτό. Θα πρέπει να δράσουμε ταχύτατα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, μέχρι το τέλος του χρόνου, κατά πάσα πιθανότητα, η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος θα είναι όνειρο απατηλό στην ε, Πολωνία. Θα πρέπει λοιπόν και στην περίπτωση της Ουγγαρίας να δράσουμε κατεπήγοντος. Και επαναλαμβάνω ότι έχουμε πολλές χώρες που έχουν παρόμοιες μεταρρυθμίσεις. Στην εμπειρία μας στην Ένωση Δικαστών, όταν κάποιος επιτίθεται στο κράτος δικαίου και στους κανόνες της δημοκρατίας, η πρώτη χειρουργική επέμβαση είναι συνήθως τα δικαστηρία, η δικαστική εξουσία. Γιατί από τον έλεγχο των δικαστών ε, μπορεί κανείς να ασκήσει έλεγχο και μετά σε πολλούς άλλους τομείς. Αυτό το έχουμε δει επανελειμμένα και έχουμε καθυστερήσει στην αντίδρασή μας έχουμε καθυστερήσει. Και γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο σημαντικό να μην γίνει διάλογος εφόσον δεν υπάρχουν και μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση, κάτι θα πρέπει να κάνουμε για να προασπιστούμε το κοινωτικό δίκαιο. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο Μάρσαλ, όπως σας είπα, για το κράτος δικαίου. Ιδάλλως το παιχνίδι θα λήξει το παιχνίδι έχει παιχθεί. Επαναλαμβάνω ότι είμαι δικαστή, είμαι τεχνικό εμπειρογνώμονα. Ναι, διακόπτει ο πρόεδρο. Αν θα μπορούσατε να ολοκληρώνετε σιγά σιγά γιατί δεν έχουμε χρόνο. Μάλιστα. Δύο προτάσει μόνο. Έλεγα ότι είμαστε εμπειρογνώμονε. Είναι τεχνική η συμβολή μα, αλλά χρειάζεται πιο ενεργής παρέμβαση και γι' αυτό Κάνουμε αυτό που κάνουμε και γι' αυτό καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η ουσία της δουλειάς μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα επιστρέφουμε στην εκπρόσωπο της Ένωσης Ιουστίτσια, της Ένωσης Πολωνών Δικαστών. Ε, σας παρακαλώ όμως να συντομεύετε και υπάρχουν και τεχνικές ε, δυσκολίες ε. με το σύστημα. Παρακαλώ. I'm sorry, is there a difficulty? Ε, συγγνώμη, υπάρχει δυσκολία να συνδεθούμε με την κυρία Χετμαρόβιτς. Είναι συνδεδεμένη. Ωραία. Με ακούτε τώρα. Ναι, ναι, έχετε τον λόγο. Για να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση για το θέμα των κυρώσεων στην κατάσταση αυτή που ζει η Πολωνία. Θα ήθελα να πω ότι ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια μέσα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να επιταχυνθούν. Αυτό πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιταχύνει την ε, διαδικασία. είναι οι διαδικασίες άτολμες και δυσκίνητες. Βλέπετε πόσο γρήγορα ε, εξελίσσεται η κατάσταση όμως στην Πολωνία. Ε, πραγματικά πολύ γρήγορα. Οπότε, επίσης θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιβάλλει την συμμόρφωση με το κράτος δικαίου. και με τις αποφάσεις του ΔΕΚ. Είναι θέμα αξιοπιστίας της Ένωσης και αρμοδιότητας ε, του ΔΕΚ επίσης. Ε, δεν μπορούμε να παριστάνουμε ότι δεν ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Οπότε πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου ε, κύρωση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτό νομίζω θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τώρα. Όσον αφορά την χρηματοδότηση των ΜΚΟ για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, νομίζω και αυτό είναι ένα μέσο το οποίο πρέπει να εξεταστεί για να απαντήσω στην δεύτερη ερώτηση. Της ε, κυρίας Ρέντκε για την ατμόσφαιρα που επικρατεί με τους δικαστές. Εδώ πέρα πρέπει να πω ότι ο νόμος αυτός, ο νόμος Φήμωτρο, όπως λέγεται, έχει κάνει πολύ κακό όσον αφορά ακριβώς το κλίμα μεταξύ των δικαστών Υπάρχει εκφοβισμός, απειλές, άλλοι απογοητεύονται. Και η πλειοψηφία των δικαστών έχει κουραστεί με την κατάσταση αυτή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν γίναμε δικαστές κανείς δεν μας προειδοποίησε ότι θα πρέπει να πολεμάμε για να υπερασπιστούμε τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το γνωρίζαμε αυτό. Υπήρχαν πολλοί δικαστές ε, που είπαν ότι δεν θα νικηθούν από τον φόβο και είναι πραγματικά πολύ γενναίοι. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε όλοι και να αναρωτηθούμε πόσο θα ε, αντέξουν. Και ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας. Πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία. Αυτό θα ήθελα να πω λοιπόν. Νομίζω ότι απάντησα στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. κύριε Χρυναλόβιτς, ευχαριστώ και τον κύριο Γκρεγραμμάτος, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που πήραν τον λόγο. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω σύντομα με κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, κάποιοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στα όσα είχε κάνει η Επιτροπή μας ε, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, το πλαίσιο κράτους δικαίου, θεμελιωδών δικαιωμάτων και δημοκρατίας με τρόπο τακτικό, περιοδικό και αντικειμενικό ε, γιατί βεβαίως αντιμετωπίζουμε τις συνήθεις ε, κατηγορίες ότι είμαστε προκατηλημένοι ε, βάσει πολιτικών πεπιθήσεων ή ιδεολογιών. Έχουμε εργαστεί λοιπόν πολύ σκληρά με βάση αυτές τις αρχές και εξετάζουμε όλα τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις συνταγματικές τους εξελίξεις, στην συμμόρφωση με τις αρχές και τις αξίες. Όπως ορίζει η συνθήκη, το άρθρο 2. Αλλά αν το Συμβούλιο ξεμπλοκάρει το αίτημα αυτό που είναι αίτημα δικό μας και της Κομισιόν για να συνδεθεί η πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια με το επίπεδο συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές αξίες, έτσι ώστε η έλλειψη συμμόρφωσης ε, να έχει δημοσιονομικές συνέπειες ε, για τις ε, χώρες που παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εάν λοιπόν οι πρωτοβουλίες αυτές αποδειχθούν αποτελεσματικές, έχουμε δουλειά μπροστά μας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα. Μας ενδιαφέρει η κατάσταση του κράτους δικαίου και θεμελιωδών ελευθεριών στην Πολωνία. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω και το έχω αναφέρει πολλές φορές. Ποτέ δεν ίσχυε ότι η δημοκρατία σημαίνει κυριαρχία της πλειοψηφίας. Βεβαίως, κυβερνάει η πλειοψηφία, ε, σύμφωνα με το κράτο δικαίου, περιοριζόμενη από το κράτο δικαίου. Η δημοκρατία δεν είναι απλά ε, η αρχή της πλειοψηφία. Περιλαμβάνει και το δικαίωμα στην αντίρρηση, την προστασία της μειοψηφίας, ε, το δικαίωμα στην αντιπολίτευση. Στο να αντιπολιτεύεται κανείς την κυβέρνηση με την ε, θεμητή βούληση τελικά να γίνει νέα πλειοψηφία και να αντικαταστήσει δημοκρατικά μέσω εκλογών την ε, εκάστοτε κυβέρνηση με μια άλλη κυβέρνηση. Οπότε η δημοκρατία δεν είναι αρχή της ε, πλειοψηφίας, είναι και η προστασία των μειονοτήτων και των δικαιωμάτων του ατόμου. Αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Αλλά υπάρχει και μια αρχή που θα ήθελα να αναφέρω Πολλέ φορέ λοιπόν έχουμε ακούσει εκπροσώπου της πολωνικής κυβέρνησης ε, στους οποίους απευθύνθηκαν πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Στον Υπουργό Δικαιοσύνη, επίσης ε, κάποια δεν απαντήθηκαν. Γι' αυτό ακριβώς ε, ζητήσαμε από τις πολωνικές αρχές να πάρουν στα σοβαρά την απόφαση, τις αποφάσεις του ε, ΔΕΚ, ε, οι οποίες είναι δεσμευτικέ για όλα τα κράτη-μέλη και για την Πολωνία και να πάρουν στα σοβαρά τις θέσεις ε, που έχει εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ψηφίσματά του, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που νομοποιείται με την άμεση ε, πλειοψηφία, με την άμεση ψηφοφορία, με συγχωρείτε, 440 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών, μεταξύ των οποίων και των 40 εκατομμυρίων Πολωνών πολιτών, που είναι Ευρωπαίοι πολίτες και έχουν κάθε δικαίωμα να ε, προστατεύονται ως Ευρωπαίοι πολίτες και να τους εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο δεν είναι ξένο, δεν είναι εξωτερική παρέμβαση στα της Πολωνίας, ε, ζητάει ε, με κάθε προσήκοντα σεβασμό από τις πολωνικές αρχές να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τις οποίες συνυπέγραψαν ε, στην συνθήκη της Λισαβόνας και να πάρουν στα σοβαρά επίσης και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις ανησυχίες μας για τα θεμελιώδη δικαιώματα και κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. και βεβαίω να ξεμπλοκάρει και το Συμβούλιο τη δικασία του άρθρου 7. Πρέπει να προχωρήσει. Ε, περάσουμε στην παράγραφο 2 και 3 του άρθρου 7. Ακόμα δεν έχουν ε, δοκιμαστεί στον δομημένο διάλογο που έχουν οι ευρωπαϊκές αρχές με τις πολιτικές αρχές. Τούτων λεχθέντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχουμε τις τροπολογίες. μέχρι τις 27 Μαΐου το μεσημέρι, 28 με το μεσημέρι. Έχουμε την ε, προθεσμία για τις τροπολογίες. Όχι, 4 το απόγευμα, τέσσερις το απόγευμα τελικά. Είναι η προθεσμία ε, υποβολής ε, τροπολογιών στο σχέδιο έκθεσης και σας ευχαριστώ για την συνεργασία. Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο κ. Κράβιτ, θέλει να μας πει κάτι. Ε, ζητώ συγγνώμη που δεν ε, είχα προσέξει ότι είστε στην αίθουσα και έχετε σχολεία. Είστε εκεί ακόμα. Ο κύριος Κραμπή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος να σας ευχαριστήσω που μας δώσατε την ε, ευκαιρία και στην ε, Ένωση Ευρωπαίων Δικαστών και ε, στην Ένωση Πολωνών Δικαστών για και να σας παρουσιάσουν το πώς έχουν τα πράγματα έτσι θα καταλάβουμε καλύτερα, καλύτερα τις ε, εξελίξεις. Είχε έρθει ο Επίτροπος στις 24 Απριλίου εδώ και σας παρουσίασε τις εξελίξεις τις τελευταίε εξελίξεις, αλλά σας είπε και το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προσιλωμένη στην υποστήριξη του κοινοτικού δικαίου και των θεμελιωδών μας ε, αξιών. Έχω να σας πω επίσης ότι από τότε, το 24 Απριλίου, είχαμε μια σειρά εξελίξεων που συνέβησαν και ξέρετε ότι αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, ξεκινήσει η διαδικασία υπερδιάσταση στις 29 Απριλίου ε, σε σχέση με αυτόν τον περιβόητο νόμο φήμοτρο και θα χρησιμοποιήσουμε ότι μας έχουμε στη διάθεσή μας ε, προς αυτή την κατεύθυνση τώρα κάτι άλλο σε σχέση με την ανάγκη για ένα νέο μηχανισμό. Όπως γνωρίζετε, εμείς ε, συντάσσουμε τώρα την έκθεση για το κράτος δικαίου του Σεπτεμβρίου. Βρίσκεται να εξελίξει η διαδικασία αυτή και θα σας ε, αναφέρομαι σχετικά οπότε πρέπει να πούμε ότι υπάρχει το κατάλληλο ρεύμα η όθηση στα πράγματα για να πάμε προς εκείνον τον μόνιμο μηχανισμό και θα έχουμε τις σχετικές αιτήσεις εκθέσεις για το κρατούς δικαίου πότε θα υπάρξει εποπτεία της κατάστασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά τις προσπάθειές σας κύριε Ισηγητά. Βέβαια εννοείται ότι είμαστε στη διάθεσή σας εάν θέλετε περαιτέρω ενημέρωση. Θα συνεργαστούμε και θα σας ενημερώνουμε. Και σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε να συμμετάσχουμε. Να είστε βέβαιος θα παρακολουθήσουμε τις ε, εξελίξεις ούτως ώστε να βοηθηθεί η υπόθεση του κοινωτικού δικαίου και των κοινωτικών αξιών. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε όλους όσους έλαβαν μέρος σε αυτήν την συζήτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστούμε και την Polsat, το πολωνικό κανάλι το οποίο μεταδίδει την ε, συνεδρίασή μας. Πάμε τώρα στο τελευταίο μας ε, θέμα, γιατί σας είπα ότι έχουμε πάντως για τις τροπολογίες μία προθεσμία. 28 Μαΐου στις 4 η ώρα. Έχουμε ακόμα λίγη ώρα και ευχαριστούμε και τους τερμινείς και την τεχνική υπηρεσία τους ευχαριστούμε γιατί θέλουμε ακόμα λίγη ωρίτσα, ούτως ώστε να μπορέσουμε σύντομα να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν σε σχέση με το τελευταίο θέμα μας οι συνάδελφοι για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Έχουμε τον εισηγητή Chris Peters. Βρίσκεται στην αίθουσα ο κύριος Peters. και θα μας ενημερώσει για την έκθεση του. Αλλά να μας ε, πούν τη γνώμη τους και οι σκιώδεις ηγητές. Κύριε Πέιτερ, έχετε το Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη τιμή που μπορούμε να σας δώσουμε πιο πολλές πληροφορίες για το περιεχόμενο της έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποβάλει ε, μια νέα νομοθεσία για την ψηφιακέ υπηρεσίε το πρώτο τέταρτο του 2020 και αναβλέθηκε αυτό στο πρώτο τρίμηνο του 2020 αναλόγω της πανδημίας του COVID ως ε, εισηγητής από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για τα θέματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ψηφιακών ε, υπηρεσιών. Καλωσορίζω αυτή τη δέσμευση που επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο ήταν μεν επιτυχή. δεν κατάφερε ωστόσο να επιλύσει το θέμα του παράνομου περιεχομένου στο διαδικτύο. Διάφορα μέλη, οι φίλοι στη Γερμανία όλο ιδιαίτερω, ενέκριναν εθνική νομοθεσία για να επιλύσουν το θέμα αυτό. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν ε, παρέμβει, θα έχουμε μια κατακαιρματισμένη αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς σαφείς κανόνες. Επίσης, έχουμε ε, χρησιμοποιήσει αρκετά πλέον αυτή την εθελούσια συνεργασία για να ξέρουμε ότι δεν αρκεί για να επιλύσουμε το θέμα του παρανόμου περιεχομένου online και χωρίς ε, περιορισμό του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης. Το θέμα λοιπόν του παράνομου περιεχομένου θα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να το επιλύσουν οι ιδιωτικέ επιχειρήσεις, πολλές εκ των οποίων δεν θέλουν καν να υπάρχει τέτοια ευθύνη και να τις βαρύνει αυτές. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσουμε γιατί μπορεί τελικά ένα είδος ε, περιεχομένου να θεωρείται παράνομο σε μια χώρα και να αποτελεί τμήμα τη προστασία των δικαιώματων στην ελευθερία τη έκφραση σε άλλο κράτο μέλο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε ότι τα εργαλεία, τα ψηφιακά που έχουμε στη διάθεσή μας δεν αρκούν για να επιλύσουν το θέμα αυτό και τελικά αυτό μπορεί να έχει αποτέλεσμα να περιοριστεί η ελευθερία έκφρασης. Από την άλλη, αν δεν χρησιμοποιηθεί ο αυτοματισμός αυτό δεν αποτελεί εναλλακτική λύση. Γι' αυτό λοιπόν σχεδόν όλες οι πλατφόρμες χρησιμοποιούν κάποιο είδους αυτοματισμό για να αντιμετωπίσουν ε, το περιεχόμενό τους. Η Facebook, για παράδειγμα, ε, ξέρετε ότι ε, αφαίρεσε 1,2 εκατομμύρια μηνύματα τα οποία είχαν ως στόχο τις χριστιανικές εκκλησίες. Είναι λοιπόν βασικό να ακολουθήσουμε τους λογαριασμούς αυτούς και διάφορα στοιχεία της, διαδικα... της οδηγίας αυτής για το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν αποδεχτεί πολύ χρήσιμα. Ως εισηγητής προτείνω να διτηρηθεί η απαγόρευση μιας γενικής υποχρέωσης εποπτείας σε ό,τι αφορά την ευθύνη για το περιεχόμενο και σε ό,τι αφορά την ιστορική αγορά για να μην υπάρχει υπερβολική συμμόρφωση και να μην υπάρχει και περιττό άχθος που να βαρύνει τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, έτσι όπως έχει το πλαίσιο σήμερα, δεν υπάρχει επαρκή διαφάνεια για τις κοινωνίες, τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών σε ό,τι αφορά το παράνομο περιεχόμενο. Επίσης, η συμπερίληψη σε αυτό το πλαίσιο δεν σημαίνει και σεβασμό των ανθρωπίνων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Χρειάζονται λοιπόν μια προσπάθεια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρξει νομική υποχρέωση για την διαφάνεια που χρειάζεται, για τις αναρμονισμένες διαδικασίες, για την ευθύνη, για το συντονισμό του περιεχομένου και ενεργά μέσα για να αποτραπεί η παρουσίαση παράνομο περιεχομένο. Έναν εξάρτητο λοιπόν σώμα θα πρέπει να δημιουργηθεί, το οποίο και θα ε, παρακολουθεί τις διαδικασίες των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών για να κάνει και ανάλυση των αλγορίθμων σε ό,τι αφορά το παράνομο περιεχόμενο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει επίσης μια τέτοια υπηρεσία την αρμοδιότητα να επιβάλλει και πρόστιμα αναλογικά όταν εντοπίζεται παράνομο ε, περιεχόμενο. Επίσης, η καλύτερη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε ότι το παράνομο περιεχόμενο θα το παρακολουθούν και οι αρχές επιβολής του νόμου. Θα πρέπει λοιπόν τέτοιο περιεχόμενο online να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια συστηματική παρακολούθηση όπως και το παράνομο περιεχόμενο άλλο. Ιδάλλως δεν θα καταφέρουμε ποτέ να έχουμε ένα δίκαιο ψηφιακό οικοσύστημα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους κλείνοντας ε, που συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή. Κλάντια Ρούμπαχ, εξαρτική δουλειά σας. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω και σε μια επικοδομητική συζήτηση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Thank you so much, Σε ευχαριστώ κύριε Πέτερς. Ε, ε, τυχερός είστε που είστε στην αίθουσα μου λένε ότι δυστυχώς έχουν απομείνει μόνο λίγα λεφτά πριν κλείσει το σύστημα. Παρακαλώ λοιπόν ισχυώδης, ένα λεπτό ο καθένας. Σοσιαλδημοκράτες. Η κυρία Μαρίνα Καλιουράντ, μπορείτε σε ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ τον κύριο Πέτερς για τη δουλειά που έκανε και τις ε, παρατηρήσεις. Και συμφωνώ με πολλά πράγματα. Ε, σε κάποια άλλα διαφωνώ. Και σε κάποια άλλα θέλω διευκρινήσεις. Και θα ήθελα να προσθέσω και κάποια άλλα σημεία με τροπολογίες, σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τον εισηγητή ότι ο γενικός στόχος ε, θα πρέπει να είναι οι χρήστες στο διαδίκτυο να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους χρήστες ε, στον αναλογικό κόσμο. Επίσης θα ήθελα να προχωρήσει η ψηφιακή ταυτοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ισχύει για όλους ε, χωρίς διακρίσεις. Θα ήθελα και εδώ πέρα συμφωνώ με τον συγητή, συμμόρφωση με την προηγούμενη νομοθεσία, το GDPR, αναφορά σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Διαφωνώ ή έχω διαφορετική άποψη για το λεγόμενο επιβλαβές ε, περιεχόμενο και θα εξηγήσω στις ε, τροπολογίες μου. Επίσης δεν συμφωνώ με την απέτηση οι πλατφόρμες να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για να κατεβάσουν το παράνομο περιεχόμενο γιατί μιλάμε για μια υποχρέωση τελικά αυτοματοποιημένων εργαλείων. Κάποια σημεία λοιπόν χρειάζεται διευκρίνηση μεταξύ των οποίων και ο νέος φορέας. Πρέπει να το συζητήσουμε και με τις άλλες ομάδες. Και τι λείπει, εγώ θα ήθελα περισσότερες αναφορές ε, στην μη διακριτική μεταχείριση και τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι η έμφαση της Επιτροπής μας. Ε, βλέπω αυτή τη στιγμή υπερβολική έμφαση στην διαχείριση του περιεχομένου. Ας περάσουμε και στα δικαιώματα και προνόμια και θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μας, γιατί ε, πρέπει οι τεχνολογίες να έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο. Στοματίσω εδώ και θα συνεργαστώ όπως είπε τον κύριο Πέτερς και τους άλλους κοιόδης συζητητές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα παρακαλώ για το Ρηνιού ο Κέρνερ έχει τον λόγο. Παρακαλώ σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ και τον κύριο Συγητή, τον κύριο Πέτερς ε, για την έκθεσή σας. Αναμένω τη συνεργασία μαζί σας. Ε. Ναι, εγώ είμαι υπέρ μιας προσέγγισης θεμελιώδων δικαιωμάτων. Πρέπει να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό το νέο καθεστώς για τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών θα είναι αναλογικό, δεν θα είναι εις βάρος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και δεν θα περιορίζει την καινοτομία, πρόσβαση πληροφορίες και την ελευθερία έκφρασης. Μην γραμμή των περισσότερων είναι ότι η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να εγγυάται το ότι υπάρχει η συμμεταχείριση οικονομικών δραστηριοτήτων online και offline ε, αρκεί να συμφωνήσουμε στην αρχή ότι θα πολεμούμε τις παράνομες δραστηριότητες με τα διανομικά δόγματα όπως κάνουμε offline. Δηλαδή προτείνω ότι οι ιδιωτικές εταιρείε δεν πρέπει να κρίνουν τι είναι νόμιμο. Αυτό ε, το κάνουν μόνο οι αρμόδιες αρχές. Δεύτερον, οι ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει στο βαθμό του δυνατού να είναι προσβάσιμες χωρίς ε, να χρειάζεται να αποκαλύψουν την ταυτότητα οι πελάτες. Οι ιδιωτικές εταιρείε δεν πρέπει να είναι υπεύθυνε για εγκλήματα που διαπράττουν οι πελάτες τους εφόσον δεν τα γνωρίζουν και δεν θα πρέπει να αναγκάζονται de jure ή de facto να επιτηρούν τους πελάτες τους για να διασφαλίσουμε ότι οι αρχές αυτές ε, δεν θα περιορίζουν την καταπολέμηση του εγκλήματος, θα πρέπει να αυξηθεί η, ε, η ικανότητα των διοκτικών αρχών. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν οι εταιρείε αυτές ε, να σέβονται τα ψηφιακά μας δικαιώματα και θα πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο υποπτίας ψηφιακών υπηρεσιών όπως γίνεται με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και κάτι οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την διαχείριση του περιεχομένου είναι οι χρήστες να έχουν μεγαλύτερη δύναμη να αποφασίζουν για το περιεχόμενο, να αποφασίζουν για την διαφήμιση και την στοχευμένη διαφήμιση. Θεωρώ λοιπόν ότι το σχετικό νομοθέτημα θα πρέπει να δώσει τον έλεγχο στους χρήστες. Σας ευχαριστώ και αναμένω την συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μπράιερ, ένα λεπτό, σας παρακαλώ, γιατί όλοι το ξεπέρασαν. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά φοβάμαι ότι το σύστημα θα κλείσει, εάν δεν σεβαστούμε τον χρόνο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Κάθε μέρα χρησιμοποιούμε τις ψηφιακέ υπηρεσίες, οπότε προτεραιότητα είναι να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και το μοντέλο είναι ο καπιταλισμός της εποπτείας. Και έχουμε επίσης και στοχευμένη διαφήμιση, έχουμε αντίστοιχες πολιτικές στις πλατφόρμες και το θέμα είναι το πώ, όπω βλέπουμε τηλεόραση, διαβάζουμε πριν τα ανώνυμα, χρησιμοποιούμε και αυτέ τι υπηρεσίε. Άρα θα πρέπει να δούμε το πώ θα, θα αντιμετωπιστεί το θέμα των αλγορίθμων του περιεχομένου, να δούμε τι θα γίνει με το αισθησιακό και ανεπιθύμητο περιεχόμενο. Να έχουμε κάποιον έλεγχο από αυτόν. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε επομένω. Θα θα γίνει με αυτά τα φίλτρα. Πολλέ φορέ τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται μπλοκάρουν του νόμιμου χρήστε πέραν του τους της ε, νοημότητας των μηνυμάτων θα πρέπει οι άρχες να μην έχουν τέτοιους ε, αναποτελεσματικούς αλγορίθμους. Να μην ισχύει η αρχή του ότι ό,τι χρησιμοποιείται εκτός ίντερνετ να χρησιμοποιείται και στο ίντερνετ. Δεν, δεν έχουμε κανένα φίλτρο όταν εγώ μιλάω ε, εκτός ίντερνετ, γιατί να έχω στο ίντερνετ. Οπότε να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις πλατφόρμες που δεν έχουν κάποιο είδους ε, διασύνδεση με κάποιες ελεκτικές υπηρεσίες και όταν έρθει η ώρα για τη σχετική τροποποίηση του κειμένου να δούμε τι θα γίνει και με το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο ίντερνετ, είχαν προτείνει οι κομισιόν Έχουμε επίσης και άλλες γνωμοδοτήσεις σχετικές που τις ετοιμάζουμε ε, και από την ΙΜΚΟ να δούμε τι έχουν να πούνε εκείνοι, τι θα πει η νομική επιτροπή. Οπότε θα συνεργαστώ με τον εισηγητή και με τους κοιόδης εισηγητές και να δω πώς θα προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή. Σας ευχαριστώ. Λέει ο κύριος Μπράιερ. Ευχαριστώ, κύριος Γιάκη από το ACR. Παρακαλώ να είστε σύντομο όμω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την έκθεση αυτή. Τι είναι το πιο σημαντικό. Φυσικά και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το έγκλημα και το έγκλημα συγκεκριμένα στο διαδίκτυο. Αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το διαδίκτυο είναι ένας χώρος όπου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται επιχειρήσεις και στον υπόλοιπο κόσμο. Άρα, αν το παρακάνουμε, θα έχουμε πολλά προβλήματα στην οικονομία μας. Άρα, αφενός προσβλέπω στη συνεργασία με τον εισηγητή προκειμένου να βρούμε νέους τρόπους να καταπολεμήσουμε το έγκλημα. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις θεμελιώδεις αξίες και ότι η ελευθερία του διαδικτύου αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για την οικονομία μας. Να δούμε λοιπόν το σύνολο της εικόνας αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος. Και τώρα να ακούσουμε και την Κορνίλια Έρνστα από την ΚΟΕ. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είναι νομίζω ένα θέμα το οποίο αξίζει τον κόμμα να το συζητήσουμε. Χαίρομαι για τη συνεργασία. Τώρα, τι θέλουμε να συζητήσουμε. Πρώτον, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τους όρους, σε ό,τι αφορά το παράνομο περιεχόμενο. Τα πράγματα δεν πέρα λίγο πιο ξεκάθαρα. Αλλά σε ό,τι αφορά το επιζήμιο αλλά μη παράνομο περιεχόμενο. Εδώ έχουμε πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον ορισμό και θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο σε ό,τι αφορά τη συζήτηση αυτή. Θα χρειαστεί κάποιο, κάποια προσαρμογή. Επίσης, σε ό,τι αφορά αυτή την ανεξάρτητη αρχεία, ακούγεται αρκετά πιστικό αυτό, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε τι σκόπο θα έχει με τέτοια υπηρεσία, να μην έχει ως σκόπο και ως αρμοδιότητα την ε, λογοκρισία με την οποία και την ε, διαφάνεια. Ύστερα, να διευκρινίσουμε ότι θέλουμε οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν διάφορα περιεχόμενα και να υπάρχουν ε, διάφορες διαδικασίες για την διαγραφή τέτοιου περιεχομένου σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, την ευθύνη. Όσο δεν γνωρίζει κανείς ότι υπάρχει το περιεχόμενο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο αν φυσικά τίθεται θέμα άρνησης να διαγράψει το περιεχόμενο εκεί είναι άλλο, άλλη υπόθεση. Είμαστε κατά των κανόνων επίσης που θα σήμαιναν περαιτέρω επιτηρήση του διαδικτύου από ιδιωτικέ εταιρείε. Τελευταίο σημείο, η παραπληροφόρηση του διαδικτύου πάντα αποτελεί ένα σημαντικό θέμα και είναι σημαντικό να δούμε πώς θα καλύψουμε καλύτερα το θέμα αυτό. Αυτά εν συντομία, εντάχει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Ένστ. Και τώρα να ακούσουμε πάλι τον κύριο Πίτερς για μια σύντομη, κάποια σύντομα σχόλια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ευχαριστώ όλους τους κοιόδης εισηγητές και αναμένω τη συνεργασία μαζί τους. Ελπίζω το στομότερο δυνατόν να μπορέσουμε να εγκρίνουμε αυτήν την έκθεση με συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πέτερς. Τα καταφέραμε. Προθεσμοί για τροπολογίες είναι 10 Ιουνίου το μεσημέρι. Αυτό έχει να πει ο πρόεδρος. 10 Ιουνίου το μεσημέρι. Και άλλη μια ανακοίνωση. Το σχέδιο γνωμοδότησης για νέα εταιρική σχέση Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκε με 52 ψήφους υπέρ 8 κατά 7 αποχές. Το σχέδιο σύστασης για δεύτερη ανάγνωση για στατιστικά στοιχεία για τη μετανάστευση και διεθνή προστασία εγκρίθηκε με 65 ψήφους υπέρ, 2 κατά και καμία αποχή. Ευχαριστούμε τους εισηγητές μας για τη δουλειά που έκαναν, το αποτέλεσμα το οποίο είναι θετικό και αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε. 4 Ιουνίου. 4 Ιουνίου. Από τις 9 το πρωί και μετά. Πρωί και απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση, για τις τεχνικές δυσκολίες που ξεπεράσαμε. Ελπίζω σύντομα να τα πούμε στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Γεια σας, με υγεία.